Um, πρέπει να ξεκινήσουμε για να μην μείνουμε πολύ πίσω στην ημερήσια διάταξη γιατί μετά θα πρέπει να φύγω και να πάω να απολαύσω την ε, διάσκεψη για τον οδικό χάρτη ή το σχεδιάγραμμα ή όπως το λέμε εν Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω στην Επιτροπή. Υποθέτω πως συγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Κανείς δεν λέει όχι. Οπότε, έγκριση των πρακτικών της 11 Απριλίου και οι τρεις συμφωνείτε. Ωραία. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Να σας πω πως ε, κατά κανόνα δεν στέλνουμε εμείς ε, αναθεωρημένη την ημερήσια διάταξη ακόμα και αν προκύψουν κάποιες αλλαγές αλλά επειδή υπήρξαν κάποιες σημαντικές αλλαγές στη σημερινή ημερήσια διάταξη θα κάνουμε μία εξαίρεση και οι βασικές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης είναι πως αναβάλλεται η έγκριση του σχεδίου ψηφίσματος για τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ και θα μετατεθεί για λίγο αργότερα σήμερα το πρωί και πάει για τις 27 Μαΐου η ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και τη στιγμή εκείνη που θα συναντούσαμε τον κύριο Επίτροπο θα συζητήσουμε την έκθεση Γκίναρ Χέκμαρτ για την ανάκαμψη πιστοτικών ιδρυμάτων η αρρύθμιση τώρα διαφέρει στην ημερήσια διάταξη από το σχέδιο που έλαβαν χτες οι βουλευτές. Φαντάζομαι βέβαια πως θα είστε όλοι μπερδεμένοι, δεν είναι και κανείς σχεδόν εντός της Αν το βλέπει κανείς από το διαδίκτυο, έτσι έχουν τα πράγματα. ορίζω τώρα τον κύριο Ρανταμάχερ, ε, Γενικό Διευθυντή της Eurostat στην ανταλλαγή αυτή απόψεων. Δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίω ήρθατε σε δύσκολη στιγμή γιατί η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα εκλογικών περιφερειών, αλλά πάρα πολλοί από τους ε, παρισταμένους βεβαίως ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της ε, στατιστικής, οπότε σας διαβεβαιώ πως μιλάτε σε ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήρθατε και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Αξιότιμοι βουλευτές, πριν από ένα χρόνο σας μίλησα για πρώτη φορά για να συζητήσουμε την κατάσταση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεσή σας να γίνει τακτική συνάντηση αυτός ο στατιστικός διάλογος γιατί έτσι αποτεικνύεται η συνειδητοποίηση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που πρέπει να έχουν οι πολιτικές σε αυτό το σημαντικό τομέα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένο από την πρόοδο που σημειώθηκε από πέρυσι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, ESS, με επικεφαλή στην Eurostat, αποδεικνύει την αξία του σε ένα δύσκολο πλαίσιο σταθερά παράγει μια ευρία κλίμακα ε, ε, επισήμων στατιστικών που είναι ουσιώδης για διάφορες πολιτικές της Ένωσης και σε εθνικά επίπεδα. Ως παράδειγμα να σας δείξω τη ροή των επισήμων στατιστικών που έχει δημοσιεύσει από αρχές Απριλίου η Eurostat. Παρακαλώ κοιτάξτε τα κείμενα που σας έχουν ε, διανεμηθεί όπου βλέπετε πόσες ανακοινώσεις τύπου έχουμε δημοσιεύσει από αρχές Απριλίου και στο μικρό ντοσχέ που σας έχει διανεμηθεί θα δείτε και μία σύντομη εκτίμηση για την, τον πληθωρισμό, το επίπεδο ανεργίας καθώς και την ανακοίνωση για το έλλειμμα και το χρέος. Και θα βρείτε και ένα μικρό φυλάδιο που είναι τριμηνιαία έκδοση που περιέχει τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία και με χαρά μπορώ να σας τα αποστέλω τακτικά για να σας βοηθήσω να έχετε πάντα τα τελευταία στοιχεία, να είστε πάντα ενημερωμένοι, αλλά μπορείτε φυσικά να τα δείτε αν ε, κατεβάσετε και ένα app στο κινητό σας από την υπηρεσία μας. Αυτό το διάγραμμα αποδεικνύει πόσο σημαντικά και αποτελεσματικά είναι αυτά τα στατιστικά στοιχεία για πολλές από τις ε, αποφάσεις σας για την πολιτική που διαμορφώνετε. Χωρίς αξιόπιστα και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, πολλές από τις ενέργειές μας θα είχαν πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης, αποτελεσματικότητας και αποδοχής από την κοινή γνώμη. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του αποδώσατε, θέτει ποσοτικούς στόχους και στατιστικές στην καρδιά της νέας οικονομικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής ε, ε, Ευρώπη 2020. Συμφωνήσαμε αυστηρές νομικές μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει ανεξαρτησία και ουσιώδης διακυβέρνηση του συστήματος αυτού. Τώρα ζητάμε να υπάρχει αποτελεσματική επιτήρηση μέσω προδιαγραφών και εργαλείων που θα μας δίνουν εγγυήσει, αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας, ακρίβειας και έγκαιρης υποβολής των δημοσιονομικών στατιστικών μας. Έχουμε κάνει σοβαρές προσπάθειες για να εξυγχρονίσουμε το κοινό σύστημα παραγωγής. Είναι ένα φιλόδοξο και μακρόπνο πρόγραμμα που θα το ακολουθήσει η Eurostat επόμενα χρόνια. Εργαζόμαστε για να διευρύνουμε την τακτική παραγωγή στατιστικών στοιχείων που θα μα επιτρέπουν, χάρη στο υψηλό επίπεδό του από πλευρά ε, ε, ουσία, ποσότητα, ποιότητα και ε, χρήση των τελευταίων επιστημονικών ανακαλύψεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε στοιχεία για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την συνοχή και την ευημερία των πολιτών. Αυτός όμως ο εξυγχρονισμός πρέπει να τύχει συνεχού υποστήριξη και ενίσχυση από τη πολιτική. Σε ορισμένε χώρε, εταίρου του συστήματο αυτού, μπορώ να σα μιλήσω σήμερα για κάποια κούραση από τι πολλέ μεταρρυθμίσεις, γιατί ήδη γίνονται βαθιές μεταρρυθμίσεις, του ζητάμε όλο και περισσότερο νέε και πιο απαιτητικέ στατιστικέ, ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλέ εξοικονομήσει ανεπαρκής πόρη. Πρέπει λοιπόν η, ε, η μεταρρυθμίσεων να είναι και σωστή και αποτελεσματική. Αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε και ποιο είναι το μέλλον του συστήματος αυτούς, αυτού. Θα μιλήσω για αυτά στο τέλος ομιλίας μου. Τώρα να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Έχουμε μια νέα προληπτική προσέγγιση τώρα, ούτω ώστε να εγγυηθούμε την ε, ποιότητα των δημοσιονομικών στατιστικών μα. Το σύστημα ενημέρωση τη 22 Απριλίου για τα ηλεκτρονικά στατιστικά στοιχεία δεν έθεσε καμία επιφύλαξη ή τροποποίηση στα εθνικά στοιχεία για δεύτερη φορά στη σειρά άλλα νέα στοιχεία. Κάθε τρίμηνο δίνουμε στοιχεία για το χρέος και το έλλειμμα των ε, κυβερνήσεων και κάθε μήνα δημοσιεύουμε αναλυτικά στοιχεία για την, ε, τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη όπου λαμβάνουμε υπόψη και την ενέργεια και τις τιμές των τροφίμων για τον πληθωρισμό. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά για σας. Η συνεργασία μας με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας συνεχίζει χωρίς ε, να υπάρξει πιστοδρόμηση παρά τις δυσχέρειες. Οι προσπάθειες αποδίδουν, σημειώνουμε ουσιώδη πρόοδο για να καταργήσουμε τις ε, παρελθούσες δυσλειτουργίες του, Ευρωπαϊκού, του ελληνικού στατιστικού συστήματος ρίζικα. Ήδη και το σύστημα ενημέρωσής μας δεν ε, έθεσε καμία επιφύλαξη για τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος της Ελλάδας για έκτη φορά στη σειρά μετά τον, ε, το φθινόπωρο του 2010. Αλλά πρέπει να υπαγρυπνούμε και να δράσουμε γιατί χρειάζεται περαιτέρω σταθεροποίηση του ελληνικού στατιστικού συστήματο. Η Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα απόφαση για την Eurostat στι 17 Σεπτεμβρίου παρελθόντο έτου, μετά την απόφαση του Προέδρου Μπαρόζο να αναθέσει τον Νοέμβριο του 2011 τη στατιστική στον Επίτροπο μέτα. Αυτό καταδεικνύει την πολιτική αποφασιστικότητα της Κομισιόν στα πλαίσια των συνθήκων για να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις και να δώσει το παράδειγμα. Η κατεξοδότηση πράξη για, τις στατιστικές, για τα στατιστικά πρόστιμα στα πλαίσια των στατιστικών ε, σε ηλεκτρονική μορφή έχει αρχίσει να ισχύει. Ανταποκριθήκαμε στο έτοιμά σας ε, στα πλαίσια του Six Pack για ε, να δράσετε κι εσείς με διαφάνεια και να συνεργαστούμε μαζί σας. Όλα αυτά βεβαίως θα απαιτήσουν πολύ χρόνο Πολύ εμπειρογνωμοσύνη και δεν θα αποτελέσουν πανάκια. Θα είναι όμως αυτή η πράξη ε, ένα όργανο ανάλογο με τις, περι, περιστάσεις. Η Eurostat σκοπεύει να ασκήσει αυτές τις νέες εξουσίες με προσοχή και ρεαλισμό. Οι διαπραγματεύσεις για το νέο εθνικό σύστημα λογαριασμών 2010, ΕΣΑ 2010 έχουν ολοκληρωθεί και ο τελικός συμβασμός περιέχει σαφή δέσμευση από πλευράς μας να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε συστηματική και επαγγελματική κάλυψη των ενδεχομένων υποχρεώσεων και να ενημερώνουμε τακτικά για αυτά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΑ 2010 από το Σεπτέμβριο 2014 όπως συμφωνήθηκε. Έχουμε μακρόπνοες φιλοδοξίες. Αρχίζουμε να προετοιμάζουμε το έδαφος για πιο συγκρίσιμες ε, στατιστικές για τα δημοσιονομικά. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει μία μελέτη σκοπιμότητας για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό ε, σύστημα ε, στατιστικών προδιαγραφών για τον δημόσιο τομέα. Έψας ε, έχουμε στόχο να συμπεριλάβουμε στοιχεία για την μέτρηση προόδου ε, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής. Πριν από μερικές μέρες προτείναμε ένα νέο σύνολο Ευρωπαϊκών οικονομικών, περιβαλλοντικών λογαριασμών, όπως είχαμε υποσχεθεί το 2011 και θα λάβετε φέτος, μία έκθεση για ε, τα στοιχεία για το ΑΕΠ και πέρα, όπως είχε ζητήσει ο, ο κανονισμός ΕΣΑ 2010. Η Eurostat παραμένει το σημείο αναφοράς για εθνικούς και διεθνείς χρήστες και από την πολιτική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την έρευνα. η ημερή αταξή μα για μεταρρυθμίσει δεν θα χαλαρώσει του επόμενου μήνε. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το στατιστικό νόμο, τον κανονισμό δηλαδή 23 223 2009. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν νέε εγγύσει για τα εθνικά στατιστικά Ινστιτούτα όσον αφορά την ανεξαρτησία του, το συντονισμό του, τι εξουσίε του και το δικαίωμα πρόσβαση σε διοικητικέ πηγέ. Επίση προτείνουμε κάθε κράτος μέλος να υπογράψει μία δέσμευση για την εμπιστευτικότητα των στατιστικών που θα είναι ένα δημόσιο πολιτικό εργαλείο που θα εγγυηθεί ότι οι προδιαγραφές στα ενωσιακά επίπεδα θα αντανακλώνται στο εθνικό επίπεδο. Οι προτάσεις μας όμως αντιμετώπισαν στεναρή αντίσταση στο Συμβούλιο. Χθες ξεκίνησαν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις και θα γίνουν πιο έντονες στις επόμενες εβδομάδες. <clears throat> Επαναλαμβάνω ότι ένας τελικός συμβασμός πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν ισότιμα αυστηρέ προδιαγραφέ και εγγυήσει σε εθνικό και ευρωπαϊκά επίπεδα. Αλλιώ θέτουμε κινδύνο το δικαίωμα και την ουσιώδη διανομή ρόλων, ευθυνών και καθηκόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματο, ούτω ώστε τα στοιχεία να παράγονται από κάτω προ τα πάνω και να από πάνω προ τα κάτω. Είμαι πεπισμένο ότι όπω και για προηγούμενε μεταρρυθμίσει, η ενεργό υποστήριξη θα μα επιτρέψει να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία και την το ρεαλισμό τη αρχική πρόταση. Πρέπει να έχουμε αρκετού πόρου για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 13-17 όταν θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για τι πολιτικες δημοσιονομικε δημοσιονομικέ προοπτικέ 2014-20. Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχία. Η Eurostat προετοιμάζει πρόταση τη Κομισιόν για έναν κανονισμό για την παροχή και ποιότητα των στατιστικών για την διαδικασία μακρο, μακροοικονομικών ανισορροπιών, MIP. Για η Eurostat είναι σαφές ότι όταν χρησιμοποιούνται οι στατιστικές ως δείκτες για σημαντικές αλλαγές πολιτικές και διοικητικές χρειάζονται ρωμαλαίες, δεσμευτικές ε, διαδικασίες επιτήρησης στη στατιστική. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν και να αποδειχθεί ότι μπορούν να επιζήσουν και των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω ε, σύντομα η Κομισιόν να εγκρίνει την πρόταση αυτή και βεβαίως θα συνεργαστούμε μαζί σας ούτω ώστε να αποφεληθούμε από τις απόψεις για την διαδικασία επιτήρηση της ποιότητα και από τη στήριξή σα για να προχωρήσει ομαλά η νομοθετική διαδικασία. Θα αναπτύξουμε τα, προαρχικα... τα προ... πρώιμα σχέδια για το έψας και θα διαπραγματευτούμε μια πρόταση για νέους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Επίσης θα αγωνιστούμε για να περάσει η πρότασή μα, για να υπάρξουν νομικέ εγγύσει για τι δημογραφικέ στατιστικέ, ούτω ώστε να είναι πλήρω συγκρίσιμε και ποιοτικά σωστέ, γιατί είναι ζωτικέ για την ε, διοργανική συζήτηση και για οικονομικέ συζητήσει όπω η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών, η πολιτική συνοχή και οι δημόσιε επενδύσει. Οι νομικέ μεταρρυθμίσει είναι αναγκαίε, αλλά όχι ικανέ. Συνεχίζουμε την ε, προσπάθειά μα για να εξυγχρονίσουμε τη διαδικασία παραγωγής και διανομής ε, στατιστικών στοιχείων. Έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, την οποία αναφέραμε στην ανακοίνωσή μας η παραγωγή στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μια, ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία που δημοσιεύσαμε το 2009. Δεν είναι εύκολο αυτό. Πρέπει να αναθεωρήσουμε 350 κανονισμούς και να μπουν σε ένα νέο πλαίσιο που θα επέτρεπε στα εθνικά στατιστικά Ινστιτούτα να αξιοποιούν πολλαπλές πηγές για στοιχεία, να μειωθούν επικαλύψεις και να υπάρξουν συνέργειες και ελαστικότητα όπως χρειάζεται. Και εδώ αντιμετωπίζουμε σημαντική προθυμία σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά την διανομή ε, στοιχείων από πηγές και τη συμφωνία επί κανόνων εμπιστευτικότητας. Επίσης, τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν πλήρως τα ευέλικτα όργανα τη ε, δευτερογενού ε, νομοθεσία που προβλέπει η Συνθήκη τη Λισαβόνα, ιδιαίτερα τη χρήση των κατεξουδότηση ε, πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 290. Είμαι πεπισμένο ότι όταν αυτό μα το όραμα γίνει πραγματικότητα, θα υποφεληθούν όλοι που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και θα μπορέσουμε να μειώσουμε τι επιπτώσει τη έλλειψη πόρων. Όπω ανέφερα προηγουμένω, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον των ευρωπαϊκών στατιστικών, πώ η ε, θεσμική δομή τους και μέθοδοι παραγωγής θα αναθεωρηθούν. Ένα νέο σύστημα ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων προκύπτει λόγω των πιεστικών αναγκών και των ε, μακρόπνων μεταρρυθμίσεων με τρεις βασικούς στόχους, ανεξαρτησία, ρωμαλαιότητα και αποτελεσματικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις μας ε, έχουν φτάσει στο όριο των νομικών δυνατοτήτων των ε, ενισχύ συνθήκων. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για ένα ουσιώδε σύστημα ευρωπαϊκών στατιστικών. Αυτή είναι η θεσμική απάντηση. Η συζήτηση αυτή θα είναι χρήσιμη, είναι επίκαιρη, ιδιαίτερα επειδή συμπίπτει με τη συζήτηση για ενδεχόμενε αλλαγέ των συνθήκων, όσο περιορισμένε και αν είναι σε αυτέ, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τη νέα οικονομική διακυβέρνηση. Έχετε υπόψη σα ότι η ΟΝΕ η νέα οικονομική διακυβέρνηση και δημιουργία πολιτικής γενικά χρειάζονται και θα μπορούσα να πω απεγνωσμένα χρειάζονται αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία. Επίσημα στατιστικά στοιχεία. Μόνιμα τονίζεται ότι οι επίσημες στατιστικές, η αξιοπιστία, ποιότητα και επάρκειά τους πρέπει να κατοχυρωθεί σαφώς και να είναι στοιχείο του πυρήνα μιας ουσιώδους ονέ. Ναι». Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας τη στήριξη. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα για την έκθεσή σας του Νοεμβρίου 2012 Προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ανέφερε τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ μεταξύ άλλων σημαντικών πολιτικών μηνυμάτων και προτεραιοτήτων. Οι σωστέ επίσημε στατιστικέ είναι βασικό εργαλείο για τρει από του τέσσερι πυλώνε, επί του οποίου μια ουσιώδη ονέ ναι πρέπει να βασιστεί. Μια επαρκή υποδομή στατιστική πληροφόρηση είναι βασική προπόθεση για τη δημιουργία και τη λειτουργία τη Δημοσιονομική Ένωση, καθώ και τη Οικονομική Ένωση. Αυτά είναι τα κλειδιά για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχει παίξει ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζω να παραμείνει και στις επόμενες συμβολές αυτής της Εμείς του Eurostat, στη Σταστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακούμε προσεκτικά τις οδηγίες και απόψεις σας. Μας έχετε βοηθήσει να αναπτύξουμε μια πολύ σημαντική ημερήσια διάταξη μεταρρυθμίσεων. Τώρα αυτό το θεματολόγιο πρέπει να είναι ακόμη πιο φιλόδοξο. Καταλήγοντας, επαναλαμβάνω ότι το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων είναι σωστό, ήδη λειτουργεί με συγκεκριμένες και ουσιώδεις ενέργειες. Τι μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία. Ότι τα επαρκή στοιχεία για σωστέ αποφάσει είναι στην καρδιά τη σωστή διακυβέρνηση. Τα στατιστικά ήταν ένα από τα πρώτα συστατικά τη δημόσια διοίκηση όταν τα ε, σύγχρονα δημόσια, ε, εθνικά κράτη δημιουργήθηκαν στην αρχή του 18ου, στο τέλος του 18ου και αρχή του 19ου αιώνα. Τώρα ζούμε σε μια περίοδο στο τέλος της οποίας το ευρωπαϊκό όραμα έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Η ιστορία μας λέει ότι οι επίσημες στατιστικές πρέπει να είναι ένα ουσιώδες τμήμα αυτής της εξέλιξης. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι σε σταυροδρόμι, όπου χρειαζόμαστε πραγματική ευρωπαϊκή στατιστική ως συμπλήρωμα μιας πραγματικής ονέ. Ναι». Το status quo δεν είναι επιλογή. Λαμβάνουμε όσο όλο και περισσότερες αιτήσει για πληροφόρηση και οι δυνατότητες ενημέρωσης ανοίγουν ευκαιρίες και ζητούν περισσότερη ευελιξία. Άρα χρειαζόμαστε ένα εξυγχρονιστικό θεματολόγιο που θεωρώ ότι είναι η κύρια αποστολή της Eurostat για τα επόμενα χρόνια. Η συνέχιση του ενδιαφέροντος και της στήριξης είναι ουσιώδης, ούτως ώστε αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και στις προσδοκίες σας. Για να βοηθήσουμε όλους τους χρήστες, όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όπως είπα και πριν, οι βουλευτές ε, εδώ πέρα <clears throat> θέλουν η Eurostat να έχει αρμοδιότητες και εξουσία γιατί βλέπουμε τα προβλήματα που προκαλούνται όταν τα ε, στατιστικά στοιχεία δεν ε, τηρούνται στο ευρωπαϊκό επίπεδο όπως θα θέλαμε. Έχω έναν κατάλογο μιλητών, οπότε ποιοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ο Σβέν σίγουρα, ο Λίαμ. Ας ξεκινήσουμε με εσά, Λίαμ. Ο Λίαμ αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται μαζί με μένα το πλαίσιο των στατιστικών στοιχείων και είναι εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου επίσης για το ΕΣΚΑΠ. Ένα πολύ δύσκολο πόστο γιατί εγώ από εκεί έγινα πρόεδρος, ο Έντγκαρ έγινε υπουργός οπότε αναφιόμαστε τι θα γίνει ο επόμενος. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Διευθυντά. Σας ευχαριστώ για την ομιλία και την παρουσίαση στόχων που κατά μεγάλο μέρος μεριζόμαστε ως προς τους φενταριστικούς στόχους και την κατάρτιση ενός σφαιρικού ολοκληρωμένου στατιστικολογικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε μεγάλη σύγκληση απόψεων και αυτό φάνηκε και από τον τριμερή διάλογο χθε. Ελπίζω λοιπόν να θα καταλήξουμε σε ευτυχές αποτέλεσμα σύντομα. Μεταξύ των δικτών που αναφέρατε ορισμένη είναι ιδιαίτερος σημαντική για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση. Ενώ τους δημοσιονομικούς δείκτες προφανώς. Παρατηρούμε σήμερα ότι ο βασικότερος αυτών των δικτών, το τρέχον δημοσιονομικό έλλειμμα, αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αρκετές χώρες αποφάσισε πλέον να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για το στόχο μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με μια διετία για τη μείωση στο 3%. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα για πολλούς αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι το να υπάρχει ένα διαρθρωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα που να είναι περιορισμένο, παρά τα μέτρα να στοχεύουν το τρέχον έλλειμμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αυτόματη σταθεροποίηση σε περιόδους ύφεση είναι ένα μεγάλο θέμα για τους αρχικού κρατών και κυβερνήσεων. Την ε, περασμένη φορά που είχατε έρθει, σα είχα θέσει μια ερώτηση για το δημοτικό αυτό έλλειμμα και μου είχατε απαντήσει και έμεινε έκπληκτος ότι δεν είχε δείκτη για αυτό το διορθωτικό έλλειμμα η Eurostat. Όμως τα περισσότερα κάτι μέλη σήμερα έχουν πλέον ε, υιοθετήσει την ε, δημοσιονομική συνθήκη, όπου ο δείκτη κλειδί για την εφαρμογή τη μακροοικονομική πολιτική είναι ακριβώ αυτό ο δείκτη του διευθυντικού ελλείμματο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. δεν πρέπει να ξεκινήσει η μελέτη αυτή ή όλη η συζήτηση για να σκεφτούμε κατά πόσον είναι εύστοχη η έννοια του διαρθρωτικού ελλείμματο, ώστε να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε την μακρονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Και σε αυτή τη φάση συλλογισμού που πρέπει να ξεκινήσει, θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για την δημιουργία αυτού του στατιστικού δείκτη, τον οποίο σας τόσο πολλοί οικονομολόγοι. Ένα σταθερό ε, μακροπρόθεσμό δείκτη που αφορά το ενδεχόμενο ποσοστό ανάπτυξης το οποίο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα εξελίσσεται, είναι αυτό που πρέπει να συγκρίνουμε με έναν βραχυπρόθεσμο διαφορετικό δίκτυο. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποια από τις δύο επιλογές είναι πιο εύστοχη, διότι οι συγκυρίες επηρεάζουν και τα διαφορετικά στοιχεία, τα δομικά. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι ακόμη και οι οικονομολόγοι δεν έχουν καταλήξει συμπερισμένα αφιλεγόμενο το θέμα. Είναι λοιπόν στην καρδιά του όλου προβληματισμού το σημείο αυτό. Δεν πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση έστω άτυπη, έστω ανεπίσημη για να αναζητήσουμε στοιχεία για το δίκτυο αυτό, γιατί πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αυτό θα βρεθεί στην καρδιά τη ερχόμενη ε, περίοδου προγραμματισμού. Για ένα, να σα δώσω ένα παράδειγμα, σε μια χώρα όπω η Γαλλία, ανάλογα με τα στατιστικολογικά ε, Ινστιτούτα, μπορεί να υπάρχουν δύο ψηφία διαφορά σε έναν δίκτυο όπω αυτό του διοικητικού ελλείμματο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αυστηροί στον καθορισμό αυτού του δίκτυου και δεν νομίζω ότι μπορεί η Eurostat να αποσιάζει από μια τέτοια συζήτηση. Well, thank uh, πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Που με κάνει να σκεφτώ τον, τους ρόλους των διαφόρων φορέων σε αυτή τη συζήτηση. Και θα επανέλθω στη διατύπωση της ερώτησής σας. Εμείς οι στρατιωτικολόγοι πρέπει να συμμετέχουμε στις συζητήσεις δικτών όποτε αυτή γίνεται σε επίπεδο πολιτικής ή έρευνας. Εμείς κατά κανόνα δεν θέλουμε να σχεδιάζουμε τους δείκτες. Παράγουμε βεβαίω στέρεα δεδομένα και πρέπει να είμαστε παρόντες όταν ε, συζητιούνται οι δείκτες, αλλά δεν είμαστε οι αρχιτέκτονες, θα έλεγα, των δείκτων. Οπότε το επανέλθω αυτό το οποίο είχα πει πέρσι. Το εάν το διαρθρωτικό έλλειμμα είναι κάτι το οποίο είναι ε, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο δίκτυ είναι ένα θέμα. Το εάν μπορεί να μετρηθεί με τρόπο αξιόπιστο είναι κάτι διαφορετικό. Η δική μου η ευθύνη αφορά το δεύτερο. Οπότε δεν θα ήθελα να δεσμευτεί η Eurostat να σχεδιάσει έναν νέο δείκτη που θα λέγεται διαρθρωτικό έλλειμμα, γιατί περιέχει αρκετά στοιχεία που είναι δύσκολα μετρήσιμα, με διάφορες ε, συμβάσεις ε, και μοντέλα, πράγματα τα οποία δεν είναι απλά για κάποια επίσημη στατιστική υπηρεσία. Αλλά αυτό το οποίο θα κάνουμε νομίζω είναι να διευρύνουμε το εύρος ε, έτσι ώστε όλα τα νομικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να γίνει κάτι τέτοιο να υπάρχουν. Ε, αν δείτε την, το δελτίο τύπου, θα δείτε, το δελτίο τύπου για το έλλειμμα και το χρέος είναι πολύ ευρύτερο και καλύπτει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν καλύπταμε πριν από 3-4 χρόνια. Ε, διάφορες λοιπόν υποχρεώσεις από εγγυήσεις ε, σε όλες τις μορφές θα συμπεριλαμβάνονται μαζί με όλους τους υπόλοιπους ε, καθορισμένους ε, δείκτες. Οπότε εμάς το βασικό μας καθήκον είναι βεβαίως να έχουμε σωστά δεδομένα για τα κριτήρια του Μάστριχτ και βεβαίως συμπεριλαμβάνουμε και άλλα στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βέρνερ. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ράντεμαχα επιβεβαιώσετε ακόμη μια φορά πως τώρα επιτέλους μετά πολλά χρόνια έχετε περισσότερες ε, αρμοδιότητες και άρα είναι πιο σημαντικά τα δεδομένα που συλλέγετε. Το ερώτημά μου είναι υπάρχει διάθεση από τις Εθνικές Αρχές για στενότερη συνεργασία ή υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Δεύτερον, ε, με φιλικό ε, τρόπο μας στείλατε αυτό το φυλάδιο με τα βασικά δεδομένα ε, στα οποία έχω κάποια ερωτήματα ως προς την ε, συγκρισιμότητα σε δύο θέματα. Το ένα αφορά το 16,9% αύξησης ε, το οποίο κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού που αναφέρατε για μια αύξηση 16,9% και 24% που αναφέρατε και το άλλο αφορά τις ε, δημοσιονομικές ε, ανισορροπίες που αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης και τέθη ήδη ένα ερώτημα για το πόσο επίκαιρα είναι τα δεδομένα σας και εάν ε, διαπιστώσατε το 2012 κάποια αλλαγή σε αυτές τις ανισορροπίες και στην Ευρώπη των 27 και στην Ευρωζώνη των 17. Okay. Let, let me... Uh, Να απαντήσω. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω πρώτα στην διάθεση συνεργασίας ε, των κρατών μελών. Όπως είπα, υπάρχουν 350 στατιστικοί κανονισμοί που καθορίζουν την θέληση αυτή. Οπότε δεν μιλάμε για το σύστημα που είχαμε στη δεκαετία του 1990 όπου ήταν θέμα επιλογής η συνεργασία, τώρα είναι νομική υποχρέωση. Είμαστε δηλαδή εντός ενός νομικού πλαισίου και οπωσδήποτε η Eurostat έχει την εξουσία να ε, εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία και να την επιβάλλει. Και αυτό γίνεται, δηλαδή ελέγχουμε την συμμόρφωση με τη στατιστική νομοθεσία για όλα τα στατιστικά στοιχεία και, και κάθε είδους. Οπότε το ζήτημα είναι του πόσο προχωράμε μετά στην επιβολή αυτής της νομοθεσίας και σε ποιο βαθμό ο νόμος ε, προβλέπει τις ε, διαδικασίες ε, παραγωγής στατιστικών στοιχείων, αλλά επί της αρχής θα έλεγα πως δεν είναι ζήτημα διάθεσης. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα είναι ένα σύστημα που βασίζεται πλέον σε νόμους και τα κράτη-μέλη κατά κανόνα συμμορφώνονται. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό της φτώχειας και την ανάπτυξη μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών. Ο πρώτος ορισμός της στόχες, για εδώ, ναι, φτώχεια μετά από τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό το δεδομένο παράγεται με συνδυασμό εθνικών λογαριασμών και κοινωνικών στατιστικών στοιχείων. Ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα κοινωνικά επιδόματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, γιατί τα συστήματα κοινωνικής αρρωγής ε, διαφέρουν, οπότε το ποσοστό της ε, φτώχειας μπορεί να υπολογιστεί μόνο αφού συνυπολογίσουμε των διαφόρων ειδών επιδόματα αλλά για το ερώτημά σας. Ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι δείκτες για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν ε, από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό μετά από τα επιδόματα. Το 16,9 είναι, θα έλεγα, το δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη ναι, αν θέλουμε να συγκρίνουμε τον κίνδυνο ε, μεταξύ κρατών μελών. Κίνδυνο για φτώχεια. Ε, όλα τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Για τον δεύτερο δίκτυ που είπατε, Εμείς ε, πρώτη φορά δημοσιεύσαμε τον, δίκ, τον κατάλογο δικτών για τον πίνακα βαθμολογίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και εδώ πέρα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επανέλθω του χρόνου όταν θα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης ε, των διαδικασιών αυτών ε, για τις ανισορροπίες γιατί Βεβαίω είμαστε στην αρχή συλλογής αυτών των δεδομένων και εδώ πέρα θα σας παραπέμψω στα συμπεράσματα τα σχετικά του Συμβουλίου για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Και ακόμη μια ερώτηση για τον κίνδυνο αυτό φτώχειας. Πώς ορίζεται, είναι ποσοστό, ε, ο ορισμός με ενδιαφέρει. Δηλαδή λέμε όποιος είναι ε, πάνω από το 50% είναι εντάξει, όποιος είναι κάτω από αυτό είναι φτωχότερος, γιατί έτσι μπορεί να γίνονται όλοι πλουσιότεροι, αλλά να παραμένει ίδιο το ποσοστό των φτωχών. Έτσι, αν γίνονται όλοι εξίσου πλούσιοι Δηλαδή έτσι είναι μόνο ένας δείκτης για την κατανομή του εισοδήματος. Αν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα, στείλτε τα γραπτός. Ε, η απάντηση. είναι έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε. Είναι ένα, ένας σχετικός δείκτης της κατανομής του εισοδήματος ε, στην κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε το μέσο εισόδημα και του νοικοκυριού και με βάση αυτό μετράμε. Αν είναι κάποιος μετά κάτω από ένα ποσοστό του μέσου εισοδήματος ε, της κοινωνίας του ε, κινδυνεύει να είναι φτωχός. Οπότε το συμπέρασμά μου είναι σωστό. Δηλαδή αυτός ο δείκτης ε, αφορά μόνο την ανισοκατανομή του εισοδήματος και όχι την πραγματική θα έλεγα φτώχεια. Ε, μιλήσατε για πραγματική φτώχεια ή απόλυτη φτώχεια. Ε, εμείς δεν μετράμε την απόλυτη ένδια. Μετράμε κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος δηλαδή είναι κάποιο ε, φτωχός, αλλά έχετε δίκιο, δεν είναι κάποια απόλυτη φτώχεια, είναι σχετική ε, εντός κάθε κράτους μέλους και κάθε κοινωνίας. Οι στατιστικές δείχνουν επίσης ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει να κάνει και με τη σχετικη ακριβώ ακριβώς φτώχεια. Πηγαίνουν πλάι-πλάι Ακόμη λοιπόν και αν είναι κανείς σχετικά πλούσιο σε μια σχετικά πλούσια χώρα, μπορεί να είναι πραγματικά αποκλεισμένο. Συγκρίνοντας αυτό το σχετικό πλούτο με τρίτες χώρες που είναι πολύ φτωχότερες. Βεν, ε, νομίζω συζήτησα στο λόγο μετά. Κατά πρώτον ευχαριστούμε που ήρθατε και για τη συζήτηση μαζί μας ένα από τα βασικά ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν είναι το κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για, τον, για την Ευρώπη του 2020. Έχουμε κάποιους βασικούς δείκτες που τους έχουμε συμφωνήσει στο Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και η Eurostat είχε δεσμευτεί στο παρελθόν να επικεντρώσει και να αφιωσιώσει πόρους στην ε, προετοιμασία και την διάθεση, διάθεση τέτοιων στοιχείων. Στον ιστότοπο σα ακόμη δεν βρίσκω βασικά δεδομένα. Όταν ε, σε ό,τι αφορά τη φτώχεια, τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα είναι από το 2010. Αυτό αποτελεί ζήτημα. Είναι πρόβλημα εάν έχετε υποσχεθεί να διαθέτετε τέτοια δεδομένα και δύο από του βασικότερου δείκτε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και απειλή από τη φτώχεια, Έχουμε διάθεση δεδομένων το 2010 τελευταία φορά. Μόλις μοιράσατε την προσούρα σας, το φυλάδιό σας, όπου εκφράζεται αισιοδοξία κατά κάποιον τρόπο, ε, γιατί βλέπω καλοκαιρινέ εικόνε εδώ και ελπίζω έτσι να παραμείνουν τα πράγματα. αισιόδοξο, όμω, στον πίνακα υπάρχει μια αρνητική υποσημείωση που δεν την καταλαβαίνω. Λέει ακριβώ κάτι για αυτά τα δεδομένα που σα είπα. Εδώ πέρα για το 2011 και 2012 τα στοιχεία για την φτώχεια και τι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κλπ. εμφανίζονται. Στην υποσημείωση τι λέει. Στην υποσημείωση, εκτός αν δεν είναι καλά τα αγγλικά μου για να καταλάβω αρκετά, ότι τα δεδομένα για το 2010 και 2011 αντικαθιστούν το 2011 και 2012 αντιστοίχω. Και το ίδιο για το 2009 και 2010 αντί για 2011-2012. Άρα, γιατί τα δεδομένα για, αυτά, για αυτούς τους βασικούς δείκτες δεν βρίσκονται στο site σας. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει εδώ κάποιος λόγος. Γιατί δεν μπορείτε να τα συγκεντρώσετε αυτά τα βασικά δεδομένα. Και τι θα κάνετε, τι θα κάνετε για να αλλάξει αυτό και μάλιστα γρήγορα. Στην ετήσια εκθεσή μας, ε, την επίσημη εκθεσή μας, για τη Eurostat έχουμε ζητήσει να γίνει πιο φιλικό προ του χρήστε το site. Δηλαδή να υπάρχουν απλέ γραφικέ παραστάσει που να μπορούν να τι δουν οι πολίτε και να τι χρησιμοποιήσουν, να τι καταλάβουν. Έκτοτε η τεχνική διάσταση του ιστοτόπου δεν έχει μεταβληθεί στο παραμικρό. Λοιπόν, πότε θα κάνετε καμιά προσπάθεια και θα υλοποιήσετε αυτά τα μέτρα να κάνετε το site τον ιστότοπο για ανθρώπους ε, που να κάνετε το site πιο ελκυστικό για ανθρώπους που θέλουν να καταλαβαίνουν τους πίνακες, λειτουργούν πιο πολύ με αυτό που πέφτει στο μάτι τους και το καταλαβαίνουν και όχι να, καταλαβαίνουν, να αναγκάζονται να καταλαβαίνουν πίνακες που μόνο οι δικοί της πληροφορικής μπορούν να αντιληφθούν. Όπως είπε ο συνάδελφος Ζαν ε, Πολ, τη μουσική των γραφικών παραστάσεων θέλουμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, Να ξεκινήσω από το τέλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε μουσική στον ιστότοπο. Δυστυχώς. Ξεκινώντας πάντως από τον ιστότοπο, από πλευρά μου να υποσχεθώ, να κάνω μια προσωπική υπόσχεση. Μικρέ αλλαγέ τι κάνουμε για να είναι το site πιο φιλικό προ το χρήστη. Προσπαθούμε να εξηγούμε τα στατιστικά στοιχεία Υπάρχει ειδικό τμήμα στον ιστότοπο που είναι φιλικό προς το χρήστη σε αυτό το ζήτημα. Είναι σαφής η γλώσσα, εξηγούνται τα πιο δύσκολα στατιστικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται πολλές γραφικές παραστάσεις και σε κάποια γωνία της οθόνης υπάρχουν και κάποια οπτικά εργαλεία όπως το ρολόι του κύκλου, του επιχειρηματικού κύκλου των ε, δικτών των τιμών και ούτω καθεξής. Τώρα, για τα υπόλοιπα τμήματα του ιστοτόπου θα χρειαστεί άλλος ένας χρόνος. Δεσμευόμαστε από τεχνικούς περιορισμούς. Όμως εγώ υπόσχομαι προσωπικά ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια. Ε, εσωτερικά γίνεται κάθε προσπάθεια να προχωρήσουμε και σας υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή την ερώτηση. Το λάβαμε το μήνυμα. Όσο για το κατά πόσον είναι επίκαιρα τα μη οικονομικά δεδομένα, όπω ρωτήσατε και εσεί, τα περιβαλλοντικά για το διοξείδιο του άνθρακα και τα κοινωνικά στατιστικά στοιχεία. Ε, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι υπάρχει καθυστέρηση στην παρουσίαση των δεδομένων αυτών. Το πρόβλημα με τη συλλογή αυτών των στοιχείων είναι ότι είναι πιο χρονοβόρα. Οι πληροφορίε που έχουμε συγκεντρώσει ω τώρα αφορούσαν περισσότερο διαθροτικά δεδομένα και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τα μεταφράσουμε σε βραχυπρόθεσμα, περισσότερο βραχυπρόθεσμα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ως προς την ενημέρωση να οδεύουν κάπως παράλληλα και με τα οικονομικά δεδομένα για το διοξίδιο του ανθρακά και για την κατανομή. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε κάποιες εκτιμήσεις φλάσσο, όπως ονομάζονται για το διοξίδιο του ανθρακά. Θα πρέπει να περιοριστούμε προ στιγμή το πώς ε, σχετίζεται το διοξείδιο του άνθρακα με την κατανάλωση ενέργειας. Έναν γενικό αριθμό για το διοξείδιο του άνθρακα που είναι όμως βασικό στοιχείο. Δεν θα ξέρουμε λεπτομέρειες για τη γεωργία και τις υπόλοιπες πηγές, όμως για την κατανάλωση ενέργειας είμαστε καθοδόν. Θα έχουμε γρήγορα κάποιες λύσεις και κάποια κοινωνικά στοιχεία. Και συνεργαζόμαστε και με αρκετά κράτη-μέλη, ιδίω αυτά που περισσότερο έχουν πληγεί από την κρίση και μαζί τους θα ετοιμάσουμε κάποιες εκτιμήσεις για την κατανομή εισοδήματο για τη διάσταση των κοινωνικών δικτών. Και πάλι λοιπόν, το λαμβάνουμε το μήνυμα, το καταγράφουμε και είμαι πεπισμένος ότι το πρόβλημα θα το λύσουμε, θα το λύσουμε στο εγγύς μέλλον για έναν επιλεγμένο αριθμό δικτών. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Εκ μέρους της ομάδας μου τη και μου Ακούσαμε τι είπατε για την υπόσχεση και την εμπιστοσύνη σας για τις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Θα κάνουμε και εμείς κάθε καλύτερη προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις ε, του τριμερούς διαλόγου και τις ερχόμενες και της προσοχής μας. Είπατε τι θα γίνει με τις υποχρεώσεις εγγυήσεων που δεν συμπίπτουν με τα κριτήρια του Μάστρικτ και δεν θα είναι διαθέσιμες στην ίδια στιγμή με, αυτά, με τα στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια του Μάστρικτ. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την πραγματική κατάσταση στην οποία βρισκόνται τα πραγματικά μέλη. Συζητούμε τι εγγύησει καταθέσεων αυτή τη στιγμή, τα σχετικά προγράμματα και την οδηγία για την ανάκτηση. Θα πρέπει περισσότερα κονδύλια να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που χρειαστεί διάθεση, διάσωση ή επίλυση μιας κατάστασης πολύ γρήγορα. Δεν έχουν βεβαίως ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις, οπότε δεν είναι σαφές ακριβώς που θα καταλήξουμε ακόμη. Όμως τελικώς φαίνεται ότι θα είναι σημαντικά τα ποσά αυτά, τα χρηματικά ποσά. Έχετε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να λογοδοτούν για αυτά τα κράτη-μέλη. Επακριβώς. Ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες στον ισολογισμό του κράτους το υπολογίζουν στο ενεργητικό. Όμως μετά τις υποχρεώσεις εγγυήσεων δεν τις βάζουν στο ίδιο τμήμα τον ισολογισμό. Είναι αυτός ένας λογικός τρόπος να επιλύεται το ζήτημα, καθότι είναι έτσι κι αλλιώς αμφιλεγόμενο. Δεν είναι σαφές ότι αυτά τα ποσά πρέπει να συσσωρεύονται με τα υπόλοιπα και να συνυπολογίζονται, τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πώς εξελίσσεται η συνεργασία γύρω στα και των των Τι έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε φέτος. Όπως είπα απαντώντας τον προηγούμενο στην πρώτη ερώτηση, θα παρατείνουμε το χρόνο ετοιμασίας δεδομένων για το έλλειμμα και το χρέος με κάποιες υποχρεώσεις για τον ισολογισμό που θα αφορούν το δοθετικό των κρατικών οργανισμών, τις υποχρεώσεις ισολογισμού των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές, τις ε, συνεργασίες ιδιωτικού δημόσιου τομέα, τα μη αποδοτικά χρέη και τη συμμετοχή των ε, κρατικών μηχανισμών σε δημόσιες επιχειρήσεις. Με το ΕΖΑ 2010, που θα είναι το νέο λογιστικό πρότυπο για τις κρατικές λειτουργίες, θα υπολογίζουμε και αυτέ τι εγγυήσει, ακόμη και αν δεν υπολογίζονται ε, στον ισολογισμό, όπω είπατε, από τα κρατη Είναι μακροσκελή ο κατάλογο και θα φροντίσουμε να σα τον ε, διαθέσουμε για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Τώρα, για το αν αυτό που είπατε ακριβώ συμπεριλαμβάνεται, δεν ξέρω, αλλά ευχαρίστω να το συμπεριλάβω, εάν ήδη δεν καλύπτεται. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο παρακαλώ. Κανένας άλλος που δεν έχει μιλήσει ακόμη. Δεν έχει μιλήσει ακόμη. Οπότε ο Σβέν μπορεί να δευτερολογήσει. Ο κύριος Γκίκολ στην έκθεση του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα ζητήσαμε να συμπεριλάβετε περισσότερα στοιχεία και να ρίξετε περισσότερο φως στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία αλληλεγγύης. Δηλαδή αυτό το τμήμα της οικονομίας που δεν είναι ούτε δημόσιο, ούτε ιδιωτικό ε, με την έννοια ότι είναι υπέρ του κέρδους, δηλαδή ε, συνεργατικές ενώσεις, ε, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όλες αυτές οι ενώσεις που για πολλούς πολίτες γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε ποιες δραστηριότητες θα αναλάβετε ε, με βάση το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος για την κατεύθυνση αυτή και επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω και για την παραοικονομία. Όταν συζητάμε θέματα για την γκρίζα ή την μαύρη παραοικονομία, βασιζόμαστε όλοι στα στοιχεία του καθηγητή Σνάιντα που τα αναφέρουν όλοι. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτά. Αν εξετάσουμε τη μεθοδολογία του, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε πολλές επικρίσεις. Θα ήθελα να μάθω εάν εξετάζεται τον τομέα αυτό, ούτω ώστε να έχουμε πιο συγκεκριμένα και επίσημα λοιπόν στοιχεία για την παραοικονομία, που είναι σημαντικό στοιχείο αυτό η παραοικονομία για τη συζήτηση που έχουμε για την φοροδιαφυγή. Ο κύριος Και τα δύο στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη συνολική μελέτη και τα στοιχεία που δίνουμε για το ΑΕΠ διότι καλύπτονται από τις δοσοληψίες ε, στις χρηματαγορές για παράδειγμα. Όλες αυτές οι συνεργατικές, μη κερδοσκοπικές ε, οργανώσεις και τα λοιπά και φορείς είναι δύσκολο να τις διαχωρίσουμε από τα συνολικά στοιχεία του ΑΕΠ. Μια ε, σκόπιμη βάση για να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις και το μέγεθος αυτού του τομέα είναι οι επισκοπήσεις για τη χρήση του χρόνου. Αυτές οι μελέτες δεν είναι συστατικό στοιχείο του κοινοτικού νομοθετικού κεκτημένου. Αλλά υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που κάνουν τέτοιες ε, μελέτες time use ε, σε τακτική δεκαετή βάση. Συζητάμε λοιπόν με τα κράτη-μέλη για να υπάρξει άλλο ένα σύνολο τέτοιων μελετών ε, time use. Συνήθως αυτές οι μελέτες γίνονται στο μέσο των περιόδων απογραφών, δηλαδή πέντε χρόνια πριν και πέντε χρόνια μετά μία απογραφή. Με αυτό έχουμε μία δυνατότητα να καταλάβουμε περισσότερο τι γίνεται για αυτές τις οργανώσεις που είναι μη κερδοσκοπικές. Η παραοικονομία τώρα. Βεβαίως. Έχουμε τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σνάιντερ. Δεν θα τις σχολιάσω. και μπορείτε να εξαγάγετε οποιοδήποτε συμπέρασμα ότι δεν είμαι διατεθειμένος ε, να τις θεωρήσω ε, ιδιαίτερα επίσημες. Ο Επίτροπός μας ε, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συλλέξουμε στοιχεία για την παραοικονομία. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ λοιπόν να δεσμευθώ ότι οπωσδήποτε θα σας χορηγήσουμε επίσημα στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά τουλάχιστον τα κράτη-μέλη που ήδη έχουν κάνει προσπάθειες για να ερευνήσουν το θέμα αυτό, είναι δετεθειμένα να συνεργαστούν μαζί μας. Οπότε ε, ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας απαντήσω καλύτερα ε, στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. ο κύριος Γκίκολτ ε, να ασχοληθώ με ε, τις απαντήσεις σας για τη δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ που ήδη ασχολείστε γιατί θα μας βοηθούσε όλους όσους διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική να έχουμε στοιχεία για αυτά. Και είναι δύσκολο σε αυτός ο τομέας, είναι γνωστό αυτό. Γιατί όποιος ε, εργάζεται στην παραοικονομία είναι δύσκολο επισήμως να μετρηθεί και οι έρευνες όμως ε, που έχουν γίνει για, για οι πανεπιστημιακές λένε ότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες στους οποίους θα μπορούσαμε να βασιστούμε. Για την πρώτη μου ερώτηση όμως, έχετε σκοπό να ασχοληθείτε συστηματικά. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της κοινωνίας των πολιτών, ίσως να ξέρετε από τη Χαϊδελβέργη, που προσπαθεί να μετρήσει τι γίνεται σε αυτήν την οικονομία της κοινωνίας και της αλληλεγγύης. Αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα και είπαν ότι πρέπει να γίνει συστηματικά η μέτρηση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλουμε να επιτύχουμε κάποια αξιοπιστία των στοιχείων. Και γι' αυτό η μελέτη της διάθεσης του χρόνου είναι ένας δείκτης. Αλλά δεν θα μπορούσαν επίσης τα κράτη-μέλη να οθηθούν να συλλέξουν χωριστά τα στοιχεία αυτών που δρούν σε διαφορετικά νομικά πλαίσια στον τομέα αυτό. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται αρκετά αξιόπιστα και γι' αυτό το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος θεωρώ ότι χρειάζεται και άλλα στοιχεία, όχι μόνο τα στοιχεία για τη μελέτη της διάθεσης του χρόνου για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό. Θα ήθελα λοιπόν να μας υποσχεθείτε ότι θα εργαστείτε περισσότερο στον τομέα αυτό. Βεβαίως ε, δεν θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, γιατί πρέπει να αλλάξει ο τρόπος για παράδειγμα, με τον οποίο τα κράτη-μέλη συλλέγουν στοιχεία για τη φορολόγηση, την απασχόληση, ούτω ώστε να έχουμε ακριβώς τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για τον τομέα αυτό. Ο κύριο Ράντερ Μάχαρ, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρω βεβαίω. Βεβαίως, ε, σκόπιμη είναι αυτή η μελέτη εδώ και χρόνια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαμε επαρκείς πόρους για να αποδώσουμε επαρκή προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Θα σας μιλήσω ανοιχτά. Νομίζω ότι οι προτεραιότητες ε, για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή, με τη θέση λειτουργία μερικών βασικών μακροοικονομικών εργαλείων. Για τους εθνικούς λογαριασμούς συγκεκριμένα. Όλοι λοιπόν οι συνάδελφοί οι συνάδελφοί μας στα κράτη-μέλη θα επενδύσουν, θα πρέπει να επενδύσουν όλες τους τις δυνατότητες ούτω ώστε μέχρι τέλους του 2014 να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για το ΕΣΑ 2010. Ίσως κατόπιν να έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε την οικονομία της κοινωνίας και της αλληλεγγύης. Τα χρόνια δηλαδή 15-17 αλλά αμφιβάλλω αν θα έχουμε επαρκές δυναμικό, επαρκές δυνατότητες. Ο κύριος Γκίγκολντ, ε, αποκαρδιωτικό αυτό. Στη χώρα μου, μετράμε το κάθε, τον κάθε λαγό που σκοτώνει ένας κυνηγό, αλλά δεν έχουμε ιδέα αν οι ενώσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς ε, δημιουργούν το 10-12% της απασχόλησης. Ο τομέας αυτός τη χάνει μεγάλης εκτίμησης ε, ε, στο ευρύ κοινό, αυτός ο τομέας της θελούσιας προσφοράς. Μετράμε κάθε είδους βλακίες, ενώ δεν μετράμε αυτά τα πράγματα που είναι τόσο σημαντικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και με ρωτάει ο μέσα αυτό πότε θα δείξουν ότι μα σέβονται μέσω τη συμπερίληψή μα στα επίσημα στοιχεία. Και αυτό που μας απαντάτε είναι ότι οι εθνικοί στατιστικοί οργανισμοί θα μετράνε το χρέος, θα μετράνε το έλλειμμά τους και δεν τους ε, ζητάει τίποτα άλλο το ΕΣΑ 2010. Ξέρω ότι είναι μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει, αλλά ειλικρινά. Σας παρακαλώ να λάβετε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα σοβαρά. Διότι εδώ αναφέρεται η σημασία που τακτικά αποδίδει το κοινοβούλιο μας σε αυτήν την οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι δευτερεύον θέμα αυτό. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, νομίζω πως πλησιάζουμε στο τέλος. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο λέει ο Σβέν, πως ε, όπως ξέρετε είμαστε τώρα σε μια διαδικασία με αρκετά κρατημέλη, όχι όλα, σε μια διαδικασία που κάποια κρατημέλη κάνουν ριζοσπαστικές αλλαγές στις ε, δαπάνες τους και βλέπουμε τα τελικά στοιχεία. Αλλά αν προσπαθήσει κανείς να έχει πιο λεπτομερείς ε, πληροφορίες για το τι είναι αποτελεσματικό και τι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, είναι δύσκολο να καταλήξουμε κάπου. Όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε αποτελεσματικοί και εάν είναι να γίνουν περικοπές να κλείνουμε προς αυτές οι οποίες έχουν λιγότερο καταστροφικά αποτελέσματα ειδικά όσον αφορά το επίπεδο φτώχειας ε, και βεβαίω ε, στην ανάπτυξη και στις θέσεις Και το να έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία από αυτά τα οποία ίσως δεν θεωρούνται δείκτες κλειδιά, νομίζω πως είναι αναγκαίο για να έχουμε ακριβώς μια πιο λεπτή αντίληψη. Έχετε κάποια σχόλια από αυτό. Ακούστε. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Βεβαίως, ακολουθούμε αυτά τα οποία μας λέτε όσο καλύτερα μπορούμε για τις προτεραιότητές μας, για το που μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας ή που μπορούμε να κάνουμε οικονομίες κάπου αλλού για να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες αλλού, αλλά δεν θα έχουμε περισσότερους πόρους είτε στο εθνικό είτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό νομίζω για την ώρα είναι ένα όνειρο μόνο. Οπότε θα πρέπει να πορευτούμε με αυτά τα οποία έχουμε. Και για να διαθέσουμε κάτι σε νέες απαιτήσεις, νομίζω χρειάζεται, όπως σας είπα, το πρόγραμμα μεταρρύθμισης του συστήματος παραγωγής στατιστικών δεδομένων. Όλα αυτά λοιπόν πάνε σε ένα νέο μεγάλο πακέτο. Αλλά νέε προτεραιότητες σημαίνει παραμέληση των ε, παλαιών. Και αυτό είναι δύσκολο βεβαίω, γιατί ε, όταν μιλάμε για τα δεδομένα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υπερασπίζονται και τα παλιά δεδομένα και τον βαθμό λεπτομέρειας που υπάρχει. Οπότε ελπίζω να αντιλαμβάνεστε πως ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ε, ε, μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο μιας λύσης ε, πακέτου. Δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο περισσότερα με τους ίδιους πόρους. Ε, αυτό θα σημαίνει, όπως σας είπα, μείωση του υπόλοιπου στατιστικού έργου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η πρόεδρος. Μπορούμε να πούμε πως ε, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα σταδιακά. Αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε για τους πόρους, βεβαίω τους περιορισμένους. Αλλά κάπως πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του αντικτύπου των μέτρων λιτότητας. Νομίζω πως έρχονται τώρα οι βουλευτές ε, και για την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Επικοδομητικός όπως πάντα και αναμένουμε την επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.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 ναι. Έχετε όλο τον κατάλογο των ε, ψηφοφοριών. Βάλτε και τις ε, κάρτες ε, στην υποδοχή. Εγώ έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Α, και όλο την ξεχνάω. Κάποιος άλλος είναι εδώ χωρίς κάρτα. Όχι, μόνο εγώ Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε ότι δουλεύουν τα μηχανήματα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Θέλετε να τελειώσουμε γρήγορα. Ψηφίστε. 9 συνάδελφοι δεν πάτησαν το κουμπί. Να ανισχύει όταν δεν μιλάτε, γιατί μπορεί κάποιος να πατάει το κουμπί και να μην ε, δουλεύει. Έχουμε τρεις, δύο ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Ένας. Ένας ακόμα. Γιατί... Μάλιστα. 33 κάρτες, 33 ψήφισαν. Ωραία. Όλοι θέλουν να τελειώσουμε γρήγορα, εκτός από δύο που δεν ξέρουν. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για την ισορροπία των φύλων ε, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Παράγραφος 1 και 2 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 3. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 6. Πέρας 15 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται Παράγραφος 5, τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 8 υπέρ. Κατά. Συγχωρείτε, τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε την τροπολογία υπέρ 8. Συν Άλλη μία βεβαίω υπέρ. Ψήφισαν όλοι, κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Κλείνει η ψηφοφορία, πέρας. 19 υπέρ, 16 κατά, δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, εποχές. Νομίζω πως είναι δεκτή, αλλά να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 9. Συν άλλη μια ψήφος υπέρ, πέρας, 20 υπέρ, 15 κατά, δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 11. Και ε, άλλη μια ψήφος βεβαίως κατά. Και άρα 17 υπέρ 18 κατά ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 8 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. και άλλη μια ψήφο να μετρήσετε κατά. Πέρας. 18 υπέρ, 17 κατά. Δεκτή. Δεν ναι, ναι, είμαστε συνεπείς νομίζω. Άρα 17 καταπίπτει. 18 η οποία είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την 18 επίσης. Άλλη μία να προσθεθεί. Πέρας. 30 υπέρ, 5 κατά. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριφθείτε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 κατά πίπτη. Παράγραφος 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Unblock μετά τα εκτιμώντας ε, α έως g υπέρ. Κατά αποχές δεκτά. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσω την τροπολογία 1 γιατί δεν είναι σαφές. 20 υπέρ, 15 κατά. Τιμώντας J υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε και αυτό. Συν άλλη μια ψήφος υπέρ. Πέρας. 17 υπέρ. 18 κατά απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο του Κάπα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Μετά αιτιολογικές αναφορές όλες μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές και περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο. Ορίστε. Μία ερώτηση για την παράγραφο 7. Οι τροπολογίες απορρίφθηκαν, αλλά δεν ψηφίσαμε το αρχικό κείμενο. Έγινε δεκτή η τροπολογία 13. Ναι, αυτή ήταν συμβατή, αλλά δεν αντικαθιστά το αρχικό κείμενο. Είναι συμβατή με το κείμενο, οπότε έχουμε το κείμενο και αυτήν μαζί. Αυτό εννοείται μάλιστα. Ναι, η 11 απορρίφθηκε, 12 απορρίφθηκε, 13 έγινε δεκτή. Μα η 13 ήταν μόνο το συμβατό μέρος. να είναι συμβατή με την παράγραφο 7 και θα ήταν συμβατή και με την με τις ε, τροπολογίες 10 και 11. Αλλά αντικαθιστά το αρχικό κείμενο. Εντάξει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε έχουμε την παράγραφο 7 συν την ε, τροπολογία 13. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα το κείμενο όπως τροποποιήθηκε Είναι άλλη μία ψήφος υπέρ. 32 υπέρ. Μία ψήφος κατά δύο εποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα παραδώσω την Προεδρία στον Πάμπλο, γιατί εγώ πρέπει να πάω στην διάσκεψη της Κομισιόν για τον Οδικό Χάρτη. anybody's against you. Morning. So good morning everyone. We move on. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο τροποποίηση πρόγραμμα τη Ένωση για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα τη χρηματοοικονομική αναφορά και του λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Στόλογιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα θυμίζω ότι η έκθεση αυτή για το πρόγραμμα 2014-2020 αφορά ένα κονδύλι των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη συγχρηματοδότηση τριών μη κυβερνητικών φορέων, οι οποίοι υποτίθεται ότι παρακολουθούν την διακυβέρνηση του διεθνούς των ε, υπευθύνων μάλλον για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που είναι οργανισμός και, το, και ο οποίο υποτίθεται ότι παρέχει συμβουλευτικέ υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λογιστικά πρότυπα. Και επίσης για την διαδικασία παροχής αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μπορεί να εγκρίνει αυτά τα διεθνή πρότυπα για την υποβολή λογιστικών εκθέσεων. Επίσης, επικεντρωνόμαστε σε θέματα διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά την, τον καθορισμό προτύπων και τον λογιστικό έλεγχο. Οι τροπολογίες που έχω προτείνει για το σχέδιο κανονισμού, όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία. Αυτά προέκυψαν από την πρώτη ανταλλαγή απόψεών μας και υπάρχει ευρεία συζήτηση σε διαφορετικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, για το θέμα ιδιαιτέρως των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μέρσταρτ που αυτή τη στιγμή είναι ειδικό σύμβουλος παρά το Επιτρόπο Μπαρνιέ και αποστολή του είναι να επικεντρωθεί στην αναθεώρηση της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών φορέων, στον τομέα της αναφοράς και των λογιστικών προτύπων, ηγείται τη συμβουλευτική ομάδα για τα λογιστικά πρότυπα, που συμβουλεύει απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επίση τη Ρυθμιστική Επιτροπή για, τη... για τα λογιστικά πρότυπα. Μια επιτροπή όπου τα κράτη-μέλη ακριβώ συζητούν τι προτάσει για τα λογιστικά πρότυπα και λαμβάνουν και αποφάσεις για το αν θα τα εγκρίνουν, θα τα επικυρώσουν αυτά τα πρότυπα ή όχι. Αυτή είναι η αποστολή, οι αρμοδιότητες του κυρίου Μέστατ. Τώρα, τι προτείνουμε με τις τροπολογίες μας. Πρώτον, να επιστήσουμε την προσοχή στη δήλωση της ομάδας του G20, διότι κάθε φορά που υπάρχει σύνοδος του G20 γίνεται μια δήλωση για την ανάγκη να υπάρξει σύγκληση σε επίπεδο διεθνών, σε επίπεδο διεθνών λογιστικών προτύπων. Δυστυχώς αυτή η πορεία προς τη σύγκληση δεν ακολουθεί καθόλου την επιθυμητή κατεύθυνση, αλλά θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις δηλώσεις που γίνονται από το G20. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή ο ειδικό σύμβουλος με στα έχει αναλάβει πλέον ε, θητεία, οπότε μια τροπολογία μας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τη βελτίωση της διακυβέρνηση αυτού του φορέως βασιζόμενη στην, ε, στις συμβουλές του ειδικού ε, συμβούλου της. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που αφορούν τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να έχει την εξουσία να, να προτείνει κατ' της πράξης, ώστε να αντικαθιστά δικαιούχο αυτού του προγράμματος συγχρηματοδότησης, εφόσον χρειάζεται, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί αυτή η αρμοδιότητα, αυτή η εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν υπάρχει ζήτημα για την επιλογή νέου δικαιούχου ή υποκατάσταση παλαιού με νέο δικαιούχο, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να υποβάλει τις ανάλογες προτάσεις. Επίσης, θέλουμε, και γι' αυτό ακριβώς προτείναμε και σχετική τροπολογία, η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, η οποία βασίζεται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε ακριβώς και σε αυτή και σε άλλες περιπτώσεις υποβολής εκθέσεων, σε κάθε τέτοιο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, να λαμβάνεται υπόψη η ακριβής μελέτη και ανάλυση των προηγούμενων προγραμμάτων ανέκαθεν επιμέναμε και μάλιστα με σαφήνεια σε αυτό το σημείο. Τώρα έχουμε αρκετές τροπολογίες που αφορούν διαφορετικές διαφορετικά καθήκοντα που θέλουμε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λόγου χάρη, λαμβάνει υπόψη προφανώς τέτοιου είδους συζητήσεις που έχουν γίνει και εδώ. Το έργο αυτών των ειδικών συμβούλων και κάποια προηγούμενα καθήκοντα που ούτως ή άλλως έφερνε εις πέραση η αλλως εφερνε Επιτροπή. Πρώτη αλλαγή που προτείνουμε είναι ο Μάρτιος του 2013 για πρώτη υποβολή έκθεσης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης για το 2014 και για τον ε, Ειδικό Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την ε, Επιτροπή τη Ρυθμιστική Επιτροπή για τα Λογιστικά Πρότυπα. Αυτή η, ε, έκθεση θα πρέπει να λάβει υπόψη τη συμβολή του Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος ούτως ή άλλως ως προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου του έχει την, ε, τον Νοέμβριο του 2013. Τον Οκτώβριο του 2014 προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια αξιολόγηση των κανονισμών για τα στατιστικά στοιχεία και τα λογιστικά πρότυπα και ενδεχομένως να υποβάλει πρόταση για την ε, αντικατάσταση την αναθεώρηση αυτών των κανονισμών. Επιπλέον, επειδή υπάρχει πρόγραμμα επταετές ούτως ή άλλως, 2014-2020, ως ήθιστε για τέτοιου είδους προγράμματα, ζητούμε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, έκθεση για το ποσοστό επίτευξης των στόχων. Υπάρχουν ακόμη δύο τροπολογίες. Η μία αφορά το δημόσιο ενδιαφέρον ακριβώς για το Συμβούλιο Παρακολούθησης το οποίο παρακολουθεί ακριβώς την όλη διαχείριση με τον σεβασμό των αρχών που πρέπει να διέπουν ε, την διαδικασία αυτή και όπως τους έχουν ορίσει αρμόδιοι για τα λογιστικά πρότυπα. Στην τροπολογία αυτή λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την ετήσια εξέλιξη στην αλλαγή της χρηματοδότησης, τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης που ε, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2013 στο προηγούμενο πρόγραμμα. Το καθήκον αυτό το, το είχαμε ούτως ή καλυπτόταν, αλλά πλέον από το 2013 μπόρεσε αυτός ο φορέας να συγκεντρώσει, να προβλέψει και άλλες πηγές χρηματοδότησης και από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι τώρα προτείνουμε αυτή την τροπολογία, η οποία αφορά όλα τα προγράμματα 2014-2020, τα οποία περιλαμβάνουν δημοσιονομικό το χαρτοφυλάκιο κρηματοδότηση και πόρους το οποίο καταγράφεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο είναι απλώς ενδεικτικό. Μέχρι να υπάρξει βέβαια συμφωνία για το πολιετες μεσονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Αυτό είναι το περιεχόμενο των τροπολογιών. Να σας πληροφορήσω ότι αύριο το πρωί θα γίνει συζήτηση συζήτηση που διοργανώνει ο κύριος Σιέρτ, ο κύριος Καμάλ μάλλον, όπου και εγώ ίδιος θα συμμετάσχω, και εκεί είναι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς χώρους, λογιστές, ακαδημαϊκοί, καθηγητές και ούτω καθεξής, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό ακριβώς των λογιστικών προτύπων. Διότι πολλά σημαντικά θέματα έχουν ε, τεθεί εδώ και εγερθεί από τους συναδέλφους στο Ευρωκοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ακριβώς τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και το πώς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτονται και απηχούνται στο έργο ακριβώς των υπευθύνων για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Είναι σημαντικό ε, και θα ήταν καλό να διοργανωθεί ίσως μια ακρόαση στο τέλος ε, του μήνα ή αργότερα. Θα δούμε ε, με τη γραμματεία πώς μπορεί να προγραμματιστεί για να καλύψουμε ακριβώς αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερως τα, πρότυπα, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ευχαριστώ κύριε Στολογιάν. Από πλευρά του σοσιαλιστή εισηγητή κύριου Αλκαντάουη, το λόγο κύριο Σάντσο Πεθέδο. Καλημέρα κύριε συνάδελφοι. Ε, Ω σκιώδη εισηγητή, ο κύριο Αλκαντάουη θέλει να ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συζήτηση αλλά ω συντονιστή στην Επιτροπή Μεταφορών έπρεπε να παρακολουθήσει μια σημαντική ψηφοφορία σήμερα το πρωί. Μου ζήτησε λοιπόν να σα διαβάσω την εξή δήλωση εκ μέρου του. Πιστεύω ότι το σχέδιο έκθεση του κυρίου Στόλογιαν οδεύει στη σωστή κατεύθυνση. Είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει να ακουστεί η ευρωπαϊκή φωνή σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αναπτυχθούν τα κατάλληλα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλου και θα πρέπει να επιταθούν οι σχετικές προσπάθειες, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει. Η συμμετοχή του κυρίου Μαϊστάτ νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επηρεάσει και το πώς θα ε, εξελιχθεί η έκθεση του κυρίου Στόλογεν σε αρκετά σημεία. Πρώτα απ' όλα το τι θα γίνει με το ε, Συμβούλιο Παρακολούθησης, όπως λέει ο κ. Μάιστατ. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ιδανική, ιδίω σε ό,τι αφορά το ρόλο και το, την αποστολή της ΕΦΡΑΓ. Κατά πρώτον, τι γίνεται με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, πώς προασπιζόμαστε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ποιος αποφασίζει τους ρόλους για δημοκρατική, τους ε, τι αρμοδιότητε για τη δημοκρατική λογοδοσία και τα λογιστικά πρότυπα των κρατών μελών και επιπλέον η, η κατάσταση για το επίπεδο IFRS, δηλαδή τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, ούτως ή άλλως δεν είναι ιδανική ακόμη. Θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς το κονδύλι 58 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί σωστά για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε σωστά και αυτού τους φορείς και το κατά πόσο ο αρμόδιος, ο σχετικός, ο ενδιαφερόμενος κλάδος θα ε, συμβάλλει. Να, να συμπεράνω λέγοντας ότι η ΦΡΑΓ θα πρέπει να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Παρακολουθήσης ώστε να υπάρξει και το πράσινο φως για να καταρτιστεί πρόγραμμα το 2014-2020 με τέτοιε συστάσει και προτάσει για μεταρρυθμίσει που θα γίνουν από τον κύριο Μάιστα αργότερα φέτο. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια μεταβατική χρηματοδότηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κλήλων, πλευρά των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και την προηγούμενη φορά Είχαμε συζητήσει αρκετά αναλυτικά την πρόταση του κυρίου Στολογιάν. Δεν έχουμε και τόσο πολλά να προσθέσουμε τώρα. Ο κύριος Μεστάτ, ε, κατά τη γνώμη μου, ε, λαμβάνει πολύ σοβαρά την αποστολή του και αυτή είναι και η βούληση του Επιτρόπου Μπαγνιέ, δηλαδή ο κύριος Μεστάτ, να μας κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Γι' αυτό διαρωτώ με τι έννοια θα είχε ε, να προχωρήσουμε και να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις χωρίς τις προτάσεις ε, του κυρίου Μεστάτ για την ε, επιχειρηματική διακυβέρνηση, για την διακυβέρνηση στον επιχειρηματικό τομέα. Θα είχε έννοια. Οι προθεσμίες λοιπόν που προτείνεται κύριε Στολογιάν είναι αρκετά φιλόδοξες. Εάν το αναβάλουμε όλο αυτό το 2014 φοβάμαι ότι δεν θα συμβούν και τόσο πολλά, γιατί όπως ξέρετε θα γίνουν ευρωεκλογές και μόνο προς το, τελ... Α, και προς το τέλος του έτους θα έχουμε και νέα επιτροπή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιδιώξουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Σίγουρα μέχρι το φθινόπωρο θα μας έχει κάνει προτάσει ο κύριος Μεστάτ. Να επιχειρήσουμε λοιπόν η όλη η επεξεργασία του θέματος της επιχειρηματικής διακυβέρνησης και του EASB ε, να αντιμετωπιστεί φέτος του οργανισμού δηλαδή για τα διεθνή ε, λογιστικά πρότυπα. Για τη χρηματοδότηση καταστήσατε σαφές ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε τελικά νούμερα γιατί δεν έχουμε ακόμη την ε, κλείσει τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ας επιχειρήσουμε να πάρουμε μόνο ένα τμήμα της χρηματοδότησης για τα πρώτα δύο χρόνια, να αποφασίσουμε γι' αυτό και να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα ε, διακυβέρνηση. Πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν αυτή η εταιρική διακυβέρνηση και ό,τι και να αποφασίσουμε να έχουμε δυνατότητα να το αναθεωρήσουμε αν αλλάξουν τα δεδομένα. Γιατί να καθορίσουμε τώρα συγκεκριμένο ποσό, νομίζω ότι θα ήταν ε, βεβιασμένο. Τελευταίο. Το ερώτημα που κυρίως μας απασχολεί, πώς θα διασφαλίσουμε την λήψη υπόψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων περισσότερο σε αυτόν τον οργανισμό ESB από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι δεν λέει επαρκή ε, στοιχεία. Δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένη η έκθεσή σας επ' αυτού. Ίσως ε, μετά τη συζήτηση που θα γίνει σε αυτή την εκδήλωση αύριο με τον Σαϊτ Καμάλ να έχουμε περισσότερα πορίσματα που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Γιατί προς στιγμήν είναι υπερβολικά γενικόλογες οι ε, απαιτήσει μας. Αν είμαστε τόσο γενικόλογοι νομίζω ότι δεν θα επιτύχουμε πολλά στην πράξη μετά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Από πλευράς των Πράσινων, ο κύριος ε, Γκίγκολ. Και κοιτάξτε, εγώ μπορώ να συμφωνήσω με αρκετά από αυτά τα οποία είπε ο Βολφ Κλίντς. Κατά την απόψή μου το βασικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί είναι πως ε, το εάν θέλουμε να στηρίξουμε τον ε, Ιεν Μάιστερτ ε, σε αυτό το οποίο κάνει. Δεν είναι σωστό να πούμε από τώρα πως ε, θα απελευθερώσουμε από τώρα τα κονδύλια. Είναι αντιφαντικό. Υπάρχουν εδώ πέρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Είχε προειδοποιήσει για κάποια πράγματα το Κοινοβούλιο στο παρελθόν, δεν είχε ακουστεί. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο Βόλφ, ότι ε, εδώ και 7 χρόνια μιλάμε για αυτή την χρηματοδότηση, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βιαστούμε υπερβολικά αλλά εκεί όπου έχουμε πραγματικά κάποια δυνατότητα επιρροής, όταν είναι δηλαδή να δώσουμε τα λεφτά, να το συνδέσουμε αυτό το θέμα με διαρθρωτικές αλλαγές. Και γιατί να βιαζόμαστε τώρα, έχετε υποβάλει την έκθεσή σας ε, κύριε Σιγητά, αλλά δεν βλέπω κάποιο λόγο να κινηθούμε τόσο γρήγορα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση πρέπει εδώ πέρα να προσκαλέσουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΦΡΑΓΟ, όπως ε, καλέσαμε και τον κύριο Μάιστερ και ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και με τον κύριο Χόγκεφόστ, έτσι ώστε αυτή η διαπραγματευτική περίοδος ε, να χρησιμοποιηθεί για να δούμε πού πάνε τα λεφτά ή αν θα ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν ή όπως λέει ο Βολφ να δούμε πρώτα θα γίνει τα δύο πρώτα χρόνια ή μια τελείως διαφορετική λύση. Να μην λίγο ανοιχτεί αυτή η υπόθεση και να εμβαθυνθεί η συζήτηση και θα πρότεινα υπό την ε, αιγίδα σας κύριε Στόλο για να προσκληθούν ο κύριος Χούγκερφος και ο πρόεδρος της ΕΦΡΑΚ για να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα για να δούμε τι γίνεται. Και να μην ε, πέσουμε στην παγίδα να απελευθερώσουμε τα χρήματα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί τα λεφτά για τα οποία μιλάμε, για το 2014 αν το δούμε, είναι πάρα πολύ ε, υψηλά αν τα συγκρίνουμε με άλλα, με τη Eurostat κτλ. Δεν ναι, υπάρχει κάποιο λόγος να σπεύσουμε εμείς να υπακούσουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν απαντάνε στα κεντρικά ερωτήματα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Με ενημερώνει η γραμματεία για να το διευκρινίσουμε. Θα γίνει μία ακρόαση εκών με τον πρόεδρο του ΕΦΡΑΓΚΑ και με τον ε, Μισελ Πράδα για να το διευκρινίσω αυτό. Από πλευρά των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος, από πλευρά του συγκεκριτή κ. Καμάλ, ο κύριος Έπη. Ευχαριστώ Πρόεδρο κύριος Καμάλ, ευχαριστώ τον συγκεκριτή για την εκθέσή του και ιδιαίτερος γιατί έχει προσκαλέσει τον κύριο Μέστατ να παραστεί σε συνεδρίαση της ΕΚΟΝ πριν από λίγες εβδομάδες τότε ε, πραγματικά ακούσαμε ποιε αρμοδιότητε έχει αναλάβει και τι περιλαμβάνει η εντολή του και τι όχι. Όπω ε, ο συγκεκριτή σημειώνει, στόχο αυτή τη Επιτροπή είναι, του Συμβουλίου είναι να ενισχύσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο κ. Καμάλ όμω δεν είναι βέβαιο ότι με περίπλοκα λογιστικά πρότυπα θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσει. Γι' αυτό θα ήθελε να οργανωθεί μια σφαιρική συζήτηση και ε, ευρύτερου πεδίου ώστε να δούμε γιατί ε, ώστε να μπορέσουν ο κύριος Τόρλογιαν και ο κύριος Καμάλ, όπως έχουν προβλέψει, αύριο στο ESP 5002 να υποδεχτούν ε, τους ομιλητές για την ακρόαση αυτή. Πρέπει να δούμε κατά πόσον θέλουμε αμερικανικό ευρωπαϊκό πρότυπο για τα λογιστικά πρότυπα και το κατά πώς μπορεί να υπάρξει σύγκληση μεταξύ πλήρως διαφορετικών συστημάτων. Ο κ. Καμάλ πιστεύει ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα λογιστικά πρότυπα έχουν φτάσει σε μια κατάσταση πραγματικής σύγχυσης. Οι επενδυτές δεν μπορούν πια να πιστέψουν τους επόπτες, ε, τους λογιστέ πολλών τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε εάν χρειάζονται και νέε δοκιμασίε ε, λεγκόπωση ε, για τι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε και προκειμένου να δούμε κατά πόσον τα λογιστικά πρότυπα αυτή τη στιγμή επαρκούν. Είναι αναγκαίε τέτοιε δοκιμέ για να δούμε κατά πόσον είναι σωστά τα πρότυπα και ο τρόπο κατάρτιση των συλλογισμών των τραπεζών. Οι προτάσει του κυρίου να οδεύουν προ αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να ενισχυθεί όλη η διαδικασία και να μην παρακολουθεί. Υπάρχουν σοβαρέ ελπίδε ότι ο κύριο Μάιστατ θα κάνει και κάποιε εύστοχε προτάσει σχετικά. Ε, η εντολή μου στον κύριο Μάιστατ θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των κυβερνητικών δομών που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται και για να υπάρξει μια σφαιρικότητα αναθεώρηση των ίδιων των προτύπων. Είναι κρίμα που η αναθεώρηση του κυρίου Μάιστατ, του κανονισμού ΑΕΣ και ε, του έργου του Συμβουλίου για τα ε, διεθνή λογιστικά πρότυπα, είναι κρίμα που όλα αυτά δεν συμπίπτουν με τους στόχους που έχουν τεθεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όμως θα πρέπει να, δούμε να θέσουμε την πρώτη θέση στι προτεραιότητέ μα την κάλυψη των αναγκών για τα λογιστικά πρότυπα. Ιδάλω, οι στόχοι μα δεν θα επιτευχθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα, να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Στην κυρία Μέλλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα όλες τις παρατηρήσεις αλλά πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα σωστού συγχρονισμού. Το αναγνωρίζουμε. Για την πρόταση αυτή, το ιδανικό θα ήταν να εγκριθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν σωστά οι δικαιούχοι, όπως εξηγείται και στην πρόταση. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή είναι ένα σημαντικό ποσοστό, 20% του προπολογισμού του ε, οργανισμού Efrag και του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όμως από το 2014 οι δικαιούχοι ακριβώς θα δυσκολεύονται. και ένα μέρος των ευρωπαϊκών λογιστικών ε, φορέων θα έχουν επίσης ε, τις χέρειες. Εάν λοιπόν οι ειδικοί σύμβουλοι δεν διευκολευθούν να καταλήγουν σε σωστές συστάσεις και αν δεν διασφαλίσουμε τα λογιστικά πρότυπα θα υπάρχει πρόβλημα. Ο κύριο Μέστα και ο συγκεκριτή σα ακριβώ αυτά τα σημαντικά ζητήματα σωστή διακυβέρνηση μελετούν, γιατί αυτά αφορούν και την ευρωπαϊκή επιρροή και την συμβολή μα και την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και ελπίζουμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά θα χρειαστεί και χρόνο για την υλοποίηση. Όπω σωστά υπογράμμισε ο κ. Καμάλ, είναι σημαντικό να δούμε τα πρότυπα αυτά καθε το περιεχόμενό του και όχι μόνο την διακυβέρνηση που σχετίζεται με τα πρότυπα αυτά. Και ακριβώ αυτή τη διάσταση, αυτή την παράμετρο, δεν την καλύπτει η θητεία του κ. του Μάιστατ. Η Επιτροπή όμως Εσωτερικής Αγοράς ακριβώς κάνει μια αξιολόγηση του σχετικού κανονισμού για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ώστε να μελετηθεί και το περιεχόμενό του. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το 2014. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να συνεξεταστούν. Διότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των ε, υπηρεσιών μα πιστεύουμε ότι αν δεν διατηρηθεί η χρηματοδότηση ω έχει τουλάχιστον το 2014, οι δικαιούχοι θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά πρότυπα. Ευχαριστώ. Να δώσω και πάλι τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Στολογιάν. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο, το μεσονομικό χαρτοφυλάκιο. Πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο με αυτό το πρόγραμμα, αλλά με όλα τα προγράμματα που για το 2014-2020 έχουν κάποιο χαρτοφυλάκιο. το θέμα αυτό το έχω ξαναθέσει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, επανειλημμένος. Τι θα γίνει εάν μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς δεν συμφωνήσουμε στο, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βάσει της συνθήκης, το 2014 θα έχουμε ένα έβδομο του δημοσιονομικού χαρτοφυλακίου που προβλέπεται για το 2014-2020, αλλά το πραγματικό πρόβλημα θα είναι οι στόχοι, οι δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται, αυτοί και αυτές θα συνεχιστούν το 2014 βάσει παλαιών προγραμμάτων και όχι βάσει των νέων ε, στοιχείων, των νέων κονδυλίων. Τέλος πάντων, δεν είναι δική μας δουλειά να, να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Είναι θέμα της Προεδρίας. Του, δικού, του, προ, του Προέδρου μας δηλαδή. Αλλά προσπαθώντας να επαναλάβω σωστά το μήνυμα που πριν από λίγες μέρες μόλις έλαβα, το Συμβούλιο δεν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για κανένα πρόγραμμα με δημοσιονομικό χαρτοφυλάκιο προτού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου προφανώς. Το ζήτημα αυτό, όπως είπα όμως, θα επιληθεί σε επίπεδο προεδριών και προέδρων. Το πώς θα εξακολουθήσουν τέτοια προγράμματα με δημοσιονομικό χαρτοφυλάκιο, με, χρηματοδότηση, θα συζητηθεί. Τώρα, η αποτίμηση της, Ευρωπα... της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους για το τι επιδιώκουμε. Εάν θέλουμε να αλλάξει το περιεχόμενο κάποιου λογιστικού προτύπου ή των λογιστικών προτύπων. Αυτό είναι ζήτημα που είναι βεβαίως ε, πολύ ενδιαφέρον για συζήτηση. Υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, προβλήματα με το περιεχόμενο των λογιστικών προτύπων. Από την άλλη όμως, πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Οι υπεύθυνοι για τα λογιστικά πρότυπα είναι ανεξάρτητοι. Οπότε προκύπτει το εξής πρόβλημα. Θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή στην κατάρτιση των λογιστικών προτύπων μέσω αυτών των φορέων που χρηματοδοτούμε. Οργανισμούς και φορείς που δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν επιρροή στο έργο των υπευθύνων για τα λογιστικά πρότυπα έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη, να γνωμοδοτήσουν. Έχουν δικαίωμα, όπως ο δικός μας οργανισμός που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προτείνουν, να παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει κάποιο λογιστικό πρότυπο, αλλά μέχρι εκεί. Άρα, πολλές συζητήσει που ήδη προαναγγέλλονται, θα γίνουν για το τα αυτά, αλλά να έχουμε και στο νου μας το εξής. Εάν σε μια διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά θέλουμε να έχουμε αποδεκτά διεθνή λογιστικά πρότυπα, αυτά τα λογιστικά πρότυπα πρέπει να καταρτιστούν από ανεξάρτητους οργανισμούς. Ιδάλλως δεν υπάρχει θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαλέξει κάποιον υπεύθυνο για τα λογιστικά πρότυπα τη αρεσκία τη και τα δικά τη λογιστικά πρότυπα, όπω τα επιλέγουν από αυτόν, να είναι όποια τη αρέσουν, αλλά να και από τα Αμερικάνικα και από τα Ιαπωνέζικα και οποιασδήποτε άλλη χώρα τα πρότυπα. Δεν είναι όμω αυτό ο στόχο ούτε του G20, ούτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε του Ευρωκοινοβουλίου, ούτε, της... ούτε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε η δυσκολία σε σχέση με την έκθεση αυτή είναι πώς να διατηρήσουμε ένα σωστό επίπεδο εξισορρόπησης της δίκαιης επιθυμία μας να μπορούμε να επηρεάσουμε το έργο της διαδικασίας δημιουργίας λογιστικών προτύπων μεν, αλλά και την προστασία ταυτόχρονα της ανεξαρτησίας των υπευθύνων για τα ίδια τα πρότυπα. σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της έκθεση αυτή. Ήδη έχω συζητήσει με τους κοιόντες εισηγητές και νομίζω έχουν δίκιο που λένε ότι αν ο ειδικό σύμβουλο Μάιστατ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του στο Νοέμβριο του 2013 και να υποβάλει στο Συμβούλιο Εκοφήν τα πορίσματα των εργασιών του, τότε, ε, λογικός, τα αποτελέσματα του έργου του πρέπει να τα δούμε και εμείς για να μπορέσουμε να τα σηματώσουμε στη δική μας την έκθεση. Οπότε εγώ δεν έχω πρόβλημα να καθυστερήσουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Αυτό παρόλα αυτά δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι των συντονιστών της Επιτροπής ΕΚΟΝ που μπορούν να αποφασίσουν σε συνάντησή τους δεν έχω πρόβλημα με την καθυστέρηση, την αναβολή. Το μέχρι πότε ας το ορίσουν στη συνάντησή τους οι συντονιστές. Διότι η έκθεση αυτή είχε ανακοινωθεί ως έκθεση προτεραιότητας μέσα σε ένα σύνολο 16 εκθέσεων που αφορούν το, διεθνές, το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Στολογιάν. Ως προ το αυστηρό πρόγραμμα, η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 23 Μαΐου, 24 μάλλον Μαΐου, αλλά θα δούμε εάν υπάρχει καμιά αλλαγή. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση συντονιστών. Η εξέταση των τροπολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις 17 Ιουνίου φέτος και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 8 Ιουλίου. Το θέμα θα περάσει από την Ολομέλεια στη Σύνοδο του Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ πολύ χρόνο, αλλά δεν βλέπω εδώ τους συζητητές. Μάλλον εδώ είναι ο εισηγητή, οπότε να περάσω στο επόμενο σημείο τη ημερήσια σε σημεία 7 και 8. Η συζήτηση θα είναι κοινή και θα εξετάσουμε σήμερα τις τροπολογίες. Στο σημείο 7 έχουμε τον κανονισμό που αφορά την αναθεώρηση των άρθρων 92-93 οριζόντες κατοικές ενισχύσεις για κάποιες περιπτώσεις μεταφορών και τον κανονισμό 994 και 98 και στο σημείο 8 τροποποίηση του κανονισμού 653-1999 του Συμβουλίου σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης. Ο λόγος πρώτα στον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίος είναι συγγητής της πρώτης έκθεσης. Δεν είναι όλοι οι σκιώδοι. Οι σκιώδεις εισηγητές εδώ, ούτε η κυρία Πιτικάινεν. Μπορεί να αλλάξει λοιπόν η σειρά με την οποία θα πάρουν οι συνάδελφοι το λόγο. Πρώτος ως να είναι ο κύριος Κούτας. Αλλά μόλις έρθει η κυρία Πιτικάινεν θα τους δώσουμε το λόγο. Κύριε ε, Ντόρφμαν. Yeah, uh... Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Έχουμε βεβαίως και τις ε, τροπολογίες ε, που κατέθεσαν οι συνάδελφοι στο εντωμεταξύ. Τις έχουμε δει και θέλω να τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική συνεργασία. Εάν δούμε το όλο ζήτημα, οι απόψεις των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων μοιάζουν σε πάρα πολλά σημεία. Θα ήθελα να είμαι σύντομος και να αναφερθώ στα σημαντικότερα σημεία. Έχουμε και κάποιες ήδη προτάσεις για συμβιβαστικές ε, τροπολογίες ε, και ε, στο να καταλήξουμε στις εξαιρέσεις, το ότι εξαιρούνται, δηλαδή ποιες κρατικές ενισχύσεις εξαιρούνται από την ειδοποίηση και να δούμε και τους διαφορούς στόχους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ο στόχος για το 2020, μετά υπάρχουν οι ερασιτέχνες αθλητές ε, ε, οι οποίοι μπορεί ταυτόχρονα βεβαίως να ασκούν και κάποια οικονομική δραστηριότητα και συμφωνούμε στο ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά την επεξεργασία αυτού του κανονισμού θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να συμμετάσχουμε και εμείς βεβαίως με στις διαδικασίες της συναπόφασης μελωδικές μελλοντικές αναθεωρήσεις. Αυτό νομίζω συμφωνούμε. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 9 της ε, πρότασης, ε, τα μαζικά μας μεταφοράς ε, και εδώ πέρα οι συνάδελφοι είναι υπέρ της εξαίρεσης από την πρόταση αυτή του Λιγότερο για ουσιαστικούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί έχουμε μια διαδικασία εδώ πέρα στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το Κοινοβούλιο στην συναπόφαση και θα θέλαμε να είναι συναπόφαση. Οπότε αν ακολουθήσουμε εδώ πέρα την πρόταση της Κομισιόν ε, αφαιρούμε αρμοδιότητες από το Κοινοβούλιο όσον αφορά δηλαδή την εξαίρεση που υπάρχει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά υπάρχει ένας άλλος υποτομέας όπου διάφοροι συνάδελφοι πρότειναν να εξαιρεθεί από την κοινοποίηση προς την ε, Κομισιόν ε, π.χ. για τον τουρισμό, ενεργειακή ασφάλεια, ε, φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, εκπαίδευση αθλητών, επαγγελματίες αθλητές, όλα αυτά σε μια συνάντηση των σχεδόν προσπαθήσαμε να τα δούμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτούς τους ε, τομείς. Αυτά λίγο πολύ από μένα, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο τον κύριο Κούτας που είναι ο σκιοδησηγητής από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για την καλή δουλειά που έχουν κάνει αλλά και για το ότι ε, επιταχύνθηκε κάπως η διαδικασία για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή πριν από το Συμβούλιο της 29ης Μαΐου. Ελπίζουμε έτσι να επηρεάσουμε την απόφαση του Συμβουλίου. Έχω υποβάλει αρκετές τροπολογίες και στις δύο εκθέσεις, μια από είμαι και στις δύο για την έκθεση Dorfman. Συμφωνώ, πρέπει να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητές μας ε, ε, στην, στο άρθρο 9 για τον 1370 του 99 για τις ε, μεταφορές ε, τις οδικές και τις ιδεοδρομικές και έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουμε την θέση του εισηγητή, δηλαδή τις τροπολογίες 38 και 56 και επίσης έχω υποβάλει και μια τροπολογία στο άρθρο 1 για να προσθεθεί ε, να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες οι κοινωνικές, οι εκπαιδευτικές και οι υπηρεσίες υγείας και επειδή ναι, λίγο, πριν την ψηφοφορία είδαμε πως ε, συμπεριλάμβανε κάποια πράγματα ο εισηγητής κάποια πράγματα οποία ζητήσαμε μετέβαλα και εγώ τη στάση μου τώρα για την εξυπηρετικά είναι βλέπουμε πως ε, είχαμε το ψήφισμα του Ιανουαρίου του 2013 όπου το Κοινοβούλιο είχε εκφράσει την άποψή του για την κοινοποίηση πληροφοριών από τους συμμετέχοντες στην αγορά, εάν οι πληροφορίες που είχαμε δεν ήταν επαρκείς. Νομίζω έτσι πως στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο, όπως εδώ πάρει, υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης έχω συντάξει κάποιες τροπολογίες που κατά την απόψή μου ενισχύουν τις κυρώσεις, δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Κομισιόν, αναφέρομαι κυρίως στην τροπολογία 33, 35 κτλ. και 38. Και βεβαίω αναμένουμε και την συνεδρίαση των σχεδόν συγητών για να δούμε τι θα γίνει με συμβαστικές λύσεις και ελπίζω και καλύτερες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χούντας. Ε, είναι εδώ η κυρία Χούντα, είναι. Α, ωραία. Να της δώσουμε το λόγο. Ως συγκήτρια για την πρώτη από τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όταν έχει κανείς δύο εκθέσεις, δύο διαφορετικές επίτροπες, ε, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Οπότε, επί της ουσίας για αυτές τις ε, κρατικές ε, ενισχύσεις, να σχολιάσω τις τροπολογίες, οι περισσότερες ε, είναι μια χαρά. Εγώ δεν υπέβαλα τροπολογίες, γιατί η Επιτροπή μας είχε υποβάλει θαυμάσιο κείμενο, είχε λάβει υπόψη τα θέματα, όπως είπα και την προηγούμενη φορά. Γενικά η προσέγγιση της Επιτροπής για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων ούτως ώστε η ίδια η Κομισιόν να ασχολείται με τις κυριότερες υποθέσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της ενιαία αγορά και βεβαίως ε, να διασφαλιστεί η σωστή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Οι τροπολογίε απλώς θέλουν να διευκρινίσουν κάποιε πλευρές της πρόταση τη Επιτροπή και γενικά είναι μια χαρά. Μια χαρά, κατά την άποψή μου. Επίσης ε, υπάρχει ενίσχυση και του ρόλου του Κοινοβουλίου και ισχυρή υποστήριξη για αυτή την ενίσχυση. Ένα νέο ρόλο του Κοινοβουλίου. Αυτό το βλέπουμε διότι στα πλαίσια των ισχυουσών συνθήκων δεν έχουμε επίσημο ρόλο στον τομέα αυτό. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο. με βάση τις υποθέσεις για τις οποίες τους ενημερώνουν οι ψηφοφόροι τους. για θέματα κατάχρησης ε, κρατικών ενισχύσεων. Οι αρμοδιότητες επιβολής ε, προστήμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων, οι τροπολογίες προτείνουν ότι θα πρέπει να είναι ανάλογες με την έκταση και φύση του υπολόγου με την έκταση και της παράβασης δηλαδή. Οι τροπολογίες 36 και 37 όπου λέγεται ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και όταν δεν συμπεριλήφθησαν αναγκαίες πληροφορίες. Καλή ιδέα. Υποστηρίζω επίσης και αυτό που ανέφερε ο συνάδελφος Έπινγκ και το ανέφερε το ανέφεραν και άλλοι ότι παρά το ότι είναι σκόπιμη αυτή η αναθεώρηση, αλλά τα δικαιώματα τρίτων και πολιτών να υποβάλουν υποθέσεις, να κάνουν προτάσεις δηλαδή για να εξεταστούν υποθέσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικά κείμενα και νομίζω ότι συμφωνεί και η Επιτροπή σε αυτό όπως βλέπετε λοιπόν. Δεν υπάρχουν ε, θεμελιώδη ζητήματα Οπότε θα προσπαθήσω να υποβάλω συμβαστικέ τροπολογίες ε, αρχέ τη επόμενη εβδομάδας και να είναι το κείμενο σαφές, να ικανοποιεί του πάντε και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Πίτη Κάινεν. Δεν βλέπω εδώ κανέναν από την Άλντε, ούτε από τους πράσινους. Οπότε, ο κύριος Έπινγκ, σκιώδης και για τις δύο εκθέσεις. Πρόεδρε, εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ούτε το Ισάλντε, ούτε των Πρασίνων, θέλω να πω τα εξή. Ε, ναι. Αφού λείπουν, προφανώ δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική ανταγωνισμού, ούτε οι πράσινοι, ούτε οι ελεύθεροι να εκφράσω τη γενική μας ανησυχία για τον εξαφανισμό των κρατικών ενισχύσεων που ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις, για τις εξαιρέσεις και για το τι συμπεριλαμβάνεται. Καταλαβαίνω την ανάγκη να υπάρξει ευθυγραμμισμός και, πλέον, και περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση. Όμως σε ό,τι αφορά τους αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό μεταξύ των αρμοδιότητων της. Μην εξαιρέσουμε υπερβολικά πολλές οικονομικές δραστηριότητες από τον έλεγχο των αρχών ανταγωνισμών ή να αποκλείσουμε αυτές που μπορεί όντω να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα κρατικών μεταφορών. Για του στόχου αυτού του κανονισμού σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να μην περιορίσουμε του επιμέρου πολίτε ε, ή να του παρατρύνουμε να υποβάλουν πολλέ προσφυγέ. Ήδη υπάρχουν δυσκολίε όμω για να εξεταστούν οι υπάρξε προσφυγέ. Μην αυξηθεί το ποσοστό του. Δεν, συμβαίνει, δεν σημαίνει επίση ότι με τον κανονισμό αυτό πρέπει να ε, πολλαπλασιάσουμε τι κατηγορίε που ήδη καλύπτονται. Ε, με πάρα πολλέ εξαιρέσει πάρα πολλού τομεί μπορεί να προκληθεί σύγχυση. Εκεί που ίσω κάποιε κατηγορίε να καλύπτονται. Θα ήταν συνετότερο να διασφαλίσουμε ότι αυτά που έχουμε και σαφή είναι και λειτουργούν ε, επαρκώς και γι' αυτό το λόγο είμαι και αντίθετο με την αυτόματη εξαίρεση από την υποχρέωση κοινοποίηση για την ε, λήψη κρατική ενίσχυση για προγράμματα ή δραστηριότητε που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκω πολύ επικίνδυνη την εικασία ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση εγγυάται την συμμόρφωση με του κανόνε των κρατικών ενισχύσεων. Αναμένω λοιπόν πραγματικά την, ε, την ε, επικοδομητική συζήτηση που θα έχουμε ακριβώ για τι συμβαστικέ τοπολογίε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε, κύριε δεν βλέπω κανέναν εκ μέρους της Γκουερτζέλ. Οπότε, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, thank you. We don't have... Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε ιδιαίτερα σχόλια. Απλώς να πούμε ότι και τα δύο θέματα συζητιούνται σήμερα το πρωί μάλιστα στο Συμβούλιο. Ενδεχομένως να είναι τελευταία συζήτηση της ομάδας εργασίας που θα λάβει υπόψη όλα τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κυρία Μέλο. Οπότε να δώσουμε πάλι το λόγο στους συγκεκριτές μας. Ο κύριος Ντόρμαν πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Οι συνάδελφοι Σκιώδης είπαν την άποψή τους, θα κάνουν μια συνάντηση τώρα των Σκιωδών και υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε ο συνάδελφος Κούτας να ψηφίσουμε ώστε να τον πιο σύντομα ούτως ώστε να επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε από αυτού την απόφαση του Συμβουλίου και ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Πιτκάινεν. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να υποβάλω συμβαστικές τροπολογίες στους σκιώδες συγητές την αρχή της επόμενης εβδομάδας και ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Πιτκάινεν. Και ευχαριστώ και τον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίος είπε, είπε ότι θα υπάρξει συζήτηση των σκιωδών στις 14 Μαΐου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Μαΐου και η έκθεση στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιούλιο. Οπότε νομίζω ότι έληξε η συνεδρίασή μας για το πρωί και θα συνεχίσουμε το σημείο 9 της ημερής της διάταξης, τον οικονομικό διάλογο με τον πρόεδρο του Eurogroup, σήμερα στις 3, στην ίδια αίθουσα. Νόμι στις 2, στις 2. Στις 2 σε αυτήν την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.